όσους δεν το άκουσαν, ότι σήμερα και πάλι ναυάγησε νοτίως της Σικελίας ένα ε, πλοίο γεμάτο πρόσφυγες που μάλλον είναι και εκατοντάδες τα θύματα που θρυνούμε. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, επαναλαμβάνονται το τελευταίο διάστημα, μήνες τώρα. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και θα φροντίσουμε τέτοιου είδου δράματα να μην ξανασυμβούν γύρω από την Ήπειρό μα. Λοιπόν,